υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου και στον πρόεδρο κ. Βαν Χομπέι. Και πάλι ήταν τιμή και χαρά για μένα το να μπορώ να εκπροσωπώ την Ιρλανδική Προεδρία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ. Έτσι λοιπόν έκλεισε η συζήτηση και ερχόμαστε τώρα στις ε, ψηφοφορίες. Καταρχήν θα ήθελα να καλέσω τον νεοεκλογέντα πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον κύριο Ονοχρή Μαλός. Σας ε, καλωσορίζουμε κύριε Μαλός. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα ε, στην μυστική ψηφοφορία για ορισμό μέλους της